που είναι το φινικέλαιο και απερίμωση και αποψήλωση των δασών. Είχαμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Σήμερα δε θα συζητήσουμε επί του σχεδίου κειμένου. Θα μας το παρουσιάσει η Κατερίνα Κονιέτσινα. Ευθύς αμέσως της δίνω το λόγο για να μας πει πώς έχουν το πράγμα, της απόψεις. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις ε, προσπάθειες ε, του σκιώδους συζητητή, θα ήθελα πραγματικά να τον ευχαριστήσω. Προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Χρειαζόμαστε μια συμβιβαστική λύση και αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για εδώ την εργασία μας στην Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης. Το θέμα των τροπικών δασών, της εξαφάνισης τους είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πιστεύω ότι με αριθμούς μπορώ να σας αποδείξω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και όσον αφορά τις επιπτώσεις σε πολύ σημαντικούς οικονομικούς τομείς, τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ε, Γραμματεία για την στήριξή της. Πρέπει επίσης να σας πω ότι εξαφανίζονται κάθε χρόνο πάρα πολύ σημαντικές ε, εκτάσεις ε, στην ε, Ινδονησία, παραδείγματο χάρη, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Είχαμε μία ακρόαση πολύ πρόσφατα και τους τελευταίους δύο μήνες πρέπει να σας πω ότι διαπιστώσαμε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Πιστεύω ότι εδώ ο ρόλος των συντονιστών ήταν καθοριστικός. Η Επιτροπή επίσης έχει συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση αυτή και ήδη από το Φεβρουάριο αυτού του χρόνου η έκθεση που έπρεπε να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την εξαφάνιση των δασών, την αποψήλωση των τροπικών δασών, ήταν ενδεχομένως για μας και ένα πρώτο βήμα πάνω στο οποίο θέλαμε να βασιστούμε. Η σύσταση 8, η σύσταση 16, το θέμα της πιστοποίησης παραδείγματος χάριν, καθώς και οι προδιαγραφές για να βασιστούμε για τις τιμές, τις κατώτατες τιμές για το 2017. Σίγουρα πιστεύω ότι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε για την πιστοποίηση θα πρέπει να γίνει πολύ πιο αυστηρό και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι θα ενσωματώσουμε και διάφορα άλλα ανησυχητικά σημεία τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε προσέξει και δεν έχουμε μπορέσει να ρυθμίσουμε. Είναι σίγουρο ότι η δική μας αξιοπιστία διακυβεύεται και θεωρώ ότι η παραγωγή φινικέλεου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για την καταστροφή αυτών των τροπικών δασών. Θεωρώ επίσης ότι και κάποιοι μικροπαραγωγοί, μικροκαλλιεργητές θα πρέπει εδώ να αποκτήσουν μεγαλύτερη στήριξη. Θεωρώ επίσης ότι όσον αφορά τις τροπολογίες θα τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και θα προσπαθήσουμε να τις ενσωματώσουμε. Θα πρέπει να βρεθούν και εναλλακτικές ε, παραγωγές όσον αφορά επίσης και τις ε, μη πιστοποιημένες ουσίες και όλα αυτά που παράγονται με φινικέλαιο, τα προϊόντα που παράγονται με φινικέλαιο χωρίς πιστοποίηση και τα βιολογικά κάψιμα τα οποία σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να μην ε, επιβαρύνουν το περιβάλλον όσο άλλα έχουν όμως, αν θέλετε για μένα, άλλες επιπτώσεις όπως αυτές που ξέρουμε σήμερα για την αποψήλωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, αυτού του είδους τα βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πριν από 15 χρόνια, περίπου το 2000-2001, γνωρίζαμε τις ε, τιμές όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπου φινικέλαιο. Το 2000-2001 ήταν 25,3 τόνοι. Σήμερα μιλάμε για τριπλάσια παραγωγή. Έχουν ξεπεράσει τα 66, τους 66 τόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι 66 εκατομμύρια τόνους. Βλέπουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό στην έκθεση αυτή να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πτυχές γιατί όταν ξεκίνησε, αν θέλετε, η παρουσίαση του θέματος αυτού του Φινικέλεου, δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν όλες αυτές οι συνέπειες. Ξέραμε ότι στην έκθεση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις θετικές προτάσεις. Προσπαθούμε να βρούμε θετικές λύσεις. Γι' αυτό και προετοιμάσαμε με αυτόν τον τρόπο την έκθεση αυτή, με σκοπό να βρεθεί συνένεση, συμφωνία και να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι όσον αφορά τη βιωσιμότητα των λύσεων που προτείνουμε οι επιχειρήσεις που βασίζονται στο φινικέλαιο και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία δεν θα πρέπει να περιοριστούν και να απομονωθούν. Γιατί εδώ μιλάμε και για την Αφρική και για τη Λατινική Αμερική, όχι μόνο για την Ινδονησία. Και είναι προφανές ότι τα ίδια ακριβώς προβλήματα προκύπτουν και εκεί και όχι μόνο στην Ασία. Η αποψήλωση είναι κάτι που μέχρι το 2020 θα πρέπει να αρχίσει να αντιστρέφεται. Γιατί αλλιώς ένα τεράστιο κομμάτι των τροπικών δασών θα πάψει να υπάρχει. Και γνωρίζουμε και όλη την ε, βιοπικιλότητα, οι ουρακοτάγκοι παραδείγματο χάρη, που θα εξαφανιστούν από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά τα τροπικά δάση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που εμπεριέχεται σε αυτήν την ε, έκθεση <clears throat> θα είναι και οι γνωμοδοτήσει των άλλων επιτροπών, Επιτροπή ε, ΔΕΒΕ. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε και να συμπληρώσουμε τις δικές μας προτάσεις με τη γνωμοδότηση των άλλων συναρμόδιων επιτροπών, οι οποίες ε, καλούνται να γνωμοδοτήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, το θέμα, γι' αυτό και θα πρέπει να ακούσουμε όλα σας τα σχόλια, όλες σας τις παρατηρήσεις, όλες τις τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλλετε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω ένα άδειο, κενό ε, κείμενο. Θα ήθελα να συμπληρώσουμε τις προτάσεις μας, να συμπληρώσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο με σκοπό το θέμα αυτό με τόσες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν ευσυνείδητο και υπεύθυνο τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε τους στόχους της χιλιετίας, όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για την συζήτηση που θα ακολουθήσει, ελπίζω. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα να αρχίσουμε τη συνήθεια διαδικασία να λάβουν τον λόγο πρώτα πρώτα και οδησίκτες από τις πολιτικές ομάδες. Αλλά λέω να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σημείωμα που μου διαβίωσε ο κύριο Τσίρι, αν δεν λάβει το λόγο. Άρα θα μιλήσω εγώ για την ε, θέση, τη θέση του. Πα με την κυρία Κονέζα, που είναι συγγήτρια και ετοίμασε αυτό το σχέδιο κειμένου για την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας που φύγει περισσότερα από τα σχετικά ζητήματα και ε, ε, εξετάζεται το κατά πόσον φταίει το φινικέλιο στην περίμορφη και αποψήλωση των δασών. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι με τροπολογίες θα κάνω κάποιες προτάσεις ούτως ώστε αυτά τα σημεία δεν έχουν περιληφθεί για να περιληφθούν. Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει ότι οι σχετικές καλλιέργειες έχουν συμβάλει στην αποψήλωση ε, πολλών ε, δασών. Και επίσης σας τονίζω το πόσο σημαντικά είναι τα συστήματα της ε, πιστοποίησης που θεωρούνται σαν μία από τις πιθανές δυνατές λύσεις γιατί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Επίσης, με αυτές τις τροπολογίες θέλω να σας προτείνω τρόπους τόσο ώστε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το έλαιο, το φινικέλαιο και να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τις ε, βλαπτικές συνέπειες αυτού του εμπορίου γιατί το φινικέλαιο είναι ένα πιστοποιημένο προϊόν, προϊόν το οποίο προέρχεται από πιστοποιημένη καλλιέργεια. Και τώρα να δώσουμε λόγο στις άλλες πολιτικές ομάδες και το λόγο έχει ο κύριος Μπράνεν από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ε, συγχαρητήρια προς τους άλλους σκιοδοσηγητές αλλά και βέβαια στην εισηγήτρια και το φινικέλαιο είναι αναντικατάστατος συστατικό των ειδών διατροφής. Γι' αυτό και είναι σοβαρές οι συνέπειες όσον πρώτη τη χρήση της γης. Χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερες γης από όσο για άλλες καλλιέργειες. Αυτό αφορά επίσης και την τη σόγια. Farming. However, Αλλά και την κράβη που χρησιμοποιεί πολύ λιγότερα ε, λιπάσματα. Ε, οπότε για τα τροπικά δάση και για το κλίμα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μηδέν αποψήλωση των δασών από αυτή την καλλιέργεια. Και επίσης να μην καλλιεργείται σε κάποια εδάφη που δεν πρέπει. Επίσης θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να δημορφώσει άποψη και να έχει επιλογή μεταξύ βιώσιμων άλλων προϊόντων και του φινικελαίου. Οπότε θα πρέπει όταν πάει να αγοράσει κάποιο προϊόν να μπορεί να δει αν υπάρχει φινικέλαιο ε, στα συστατικά. Αναφέρεται ότι μέχρι 45-50% του φενικελαίου που εισάγεται καταλήγει στα βιοκαύσιμα και στις ζωοτροφές. Και έτσι αντισταθμίζονται όλα τα θετικά των βιοκαυσίμων. Άρα θα πρέπει να σταματήσει αυτή η χρήση. Δεν είναι βιώσιμη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε στις αναπτυσσόμενες χώρες το πόσο επηρεάζεται η χρήση της γης, αλλά και τα εμπράγματα δικαιώματα, ιδίως των μικροκαλλιεργητών και των ηθαγενών. Η παραγωγή του προϊόντος αυτού φύγει και το περιβάλλον, αλλά και την κυριότητα αυτών των γιών όπου ε, καλλιεργείται. Ο πρόεδρος. Καμία φορά θα πρέπει να επενθούμε στους Άγγλους συναδελφούς για να τους παρακαλέσουμε να μιλούν πιο αργά όταν λάβουν τον λόγο. Κύριε Γκέρλινγκ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω πολύ αργά. Όχι, εντάξει, κανονικά θα μιλήσω. Και ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την κυρία Κονέτσκα για την έκθεσή της. Και το λέω ειλικρινά ότι πιστεύω πως είναι πολύ καλά ισορροπημένη η έκθεση, γιατί έχει αποφύγει τις εύκολες ε, λύσεις ε, λαϊκισμού για να τα πει ότι όλα είναι κακά για το φινικελό έχει είναι καλά ισορροπημένη η έκθεσή της. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπράνεν που αναφέρει τα θετικά όσον αφορά το φινικέλο. Δεν θα τα επαναλάβω μια που τα είπε εκείνος. Όμως, είναι ένα μεγάλο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε και χαίρομαι που η ομάδα μου έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτή τη συζήτηση. Στις ε, αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα από πού έχουμε τα στατιστικά μας δεδομένα γιατί μερικά μπορεί κανείς εύκολα να αντιπαραλάβει, παραβάλει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σκιώδεις μεταξύ μας. Γενικότερα τώρα, συμφωνώ για τόσο αναφέρονται όσον αφορά τη συλλογική ευθύνη και αυτό θέλω να το υπογραμμίσουμε. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για δράσεις από πλευρά των χωρών που παράγουν, αλλά και από τις χώρες οι οποίες καταναλώνουν ίσως σε θελοντική βάση, όχι με νομοθεσία, αλλά θα πρέπει και αυτές να αναλάβουν μέρος της ευθύνης. Συμφωνώ για το είπε ο κ. Μπράνεν για την αποψήλωση. Αλλά επειδή παρακολούθησα τις συζητήσεις για τα βιοκαύσιμα, δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι πριν το 2020 θέλουμε να έχουμε ένα ποσοστό βιοκαυσίμων από φινικέλαιο. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που είναι ολοφάνερο είναι ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειαζόμαστε κάτι όσον αφορά τα βιοκαύσιμα για μετά το 2020. Και τι θα γίνει με το μέλλον του φινικέλου μέσα σε αυτό το μείγμα. Εδώ, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει κάτι. Η Κατερίνα καλά καταλαβαίνει τις διαφορές που υπάρχουν στα διάφορα επίπεδα πιστοποίησης και την ε, συμμόρφωση προς αυτά. Συμφωνώ μαζί της για το ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία ενιαία αναγνωρισμένη πιστοποίηση, ώστε ο κόσμος να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι όταν αγοράζει φινικέλαιο είναι από βιώσιμη παραγωγή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό 100% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως πρέπει να το προσπαθήσουμε και να το λέει αυτό η έκθεση. Σε ε, τέτοιε εκθέσει πρωτοβουλία δεν νομίζω ότι πρέπει να λέμε ότι αυτό το 100% πρέπει να το πετύχουμε τότε με ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε πω θέλουμε η τάση να είναι αυτή. Αυτό θέλουν και οι καταναλωτέ. Και τώρα για τι δυσκολίε όσον αφορά τι ετικέτε. Όντω πρέπει να προσαρμοστούμε με τόσα ισχύουν μέχρι τώρα για τους καταναλωτές Εντάξει, σίγουρα όλοι θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε 100% από βιώσιμη παραγωγή φινικέλο. Και κάτι τελευταίο, όταν μιλάμε για την αποψήλωση, δεν έχουμε πραγματικά ορισμό, δεν υπάρχει διεθνής ορισμός της αποψήλωσης. Θα ήταν χρήσιμο όμως να το προσπαθήσουμε και να το βούμε αυτό στην ε, εκθεσή μας, ιδίως όταν μιλάμε για τη Μαλισσία και την Ινδονησία που δεν έχουν εκτιματολόγιο όπως έχουμε εμείς εδώ. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών που είναι διαθέσιμα. Οπότε ας κοιτάξουμε λίγο το θέμα του ορισμού της αποψήλωσης. Γενικά πάντως πιστεύω ότι είναι μια καλή έκθεση. Θα έχω πολλές τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι θετικές, που θα ενισχύσουν την έκθεση, δεν θα πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ και πάλι την Κατερίνα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, η κυρία Ντονμάνα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όσους πήραν το λόγο και κυρίως την εισηγήτρια για το εξαίρετο έργο της. Η καλλιέργεια του φοινικέλεου σημαίνει ότι δικηδεύονται πολλά πράγματα. Αλλά χρειάζεται και μια ισορροπημένη και μετρημένη απάντηση δεν ε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι το φινικέλαιο είναι ο μόνος υπεύθυνο για την ε, αποψήλωση ή για τα αίρια του θερμοκηπίου. 50% της ε, παγκόσμιας παραγωγής 2010-2012 δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φινικέλαιο. Σίγουρα η αποψήλωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταγγείλουμε. Επίσης, από τις άλλες παραγωγές φυτικού ελαίου, το φινικέλαιο είναι αυτό που απαιτεί το, τη μικρότερη έκταση. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει μικρούς παραγωγούς, που είναι υπεύθυνοι για το 40% της παραγωγής και στρέφονται προς την παραγωγή αυτή, επειδή δεν υπάρχει άλλη παραγωγή που να τους αποδίδει τα ίδια. Και συχνά βρίσκονται σε δύσκολη θέση σε σχέση με μεγάλες ε, ομάδες που κυνηγάνε την πιστοποίηση και μάλιστα σε μια αγορά που είναι όλιγο πώλησης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν όλες τις προβληματικές που έχουν να κάνουν με το φινικέλο και να μετρήσουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης υποκατάστασης του προϊόντος αυτού. Τέλος, θέλουμε να συμφιλιώσουμε τις ανάγκες ε, τις διατροφικές και τις ενεργειακές με την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η τρίτη αγορά για το φινικέλαιο χρησιμοποιεί και για καύσιμα. 46% του φινικέλαιου καταναλώνεται στην Ευρώπη. Κανένα όμως ε, δεν προσφέρει τέτοια απόδοση όπως προσφέρει το φινικέλαιο. Οπότε αλλού για άλλε καλλιέργειε μπορεί να χρειαζόμαστε μεγαλύτερε εκτάσει. Δεν υπάρχει και άλλη καλή λύση ούτε για τι διατροφικέ μας ανάγκε. Οπότε οι βλάβες από το φινικέλαιο δεν βλέπω να είναι μεγαλύτερε από τι βλάβε από άλλα υποκατάστατα. Τα λιπαρόξα για παράδειγμα αυτό το έδειξαν. Στα πλαίσια του έργου μας, λοιπόν, καλό είναι να κρατήσουμε μια μετρημένη κατευθυντήρια γραμμή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, κύριε Μελιούρ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως κάποια από τα θέματα που θίγονται εδώ θα συμπεριληφθούν και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας που έτσι και αλλιώς θα συζητηθεί. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε δύο σημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του φινικέλαιου και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις οικονομικές επιπτώσεις και θέματα δημόσιας υγείας όπως τα τρανς λιπαρά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι ουσίες αυτές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικατασταθούν αυτά τα τρανς λιπαρά. Το φινικέλαιο βεβαίως μπορεί να βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές όπως ε, ακούσαμε για να έχουν ένα, μια πολύ καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές τους. Τέσσερις φορές καλύτερη, αν θέλετε, απόδοση από άλλες αντίστοιχες καλλιέργειες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε χρησιμοποιείται λιγότερη επιφάνεια για πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Ευχαριστώ πραγματικά την εισηγήτρια, ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές και θα ήθελα να πω ότι όλες αυτές οι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που ακούγονται θα πρέπει να ενσωματωθούν με μία κύρια ιδέα, την βιωσιμότητα τις ε, βιώσιμες καλλιέργειες και παραγωγές και πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτού του είδους τη γεωργία και αυτού του είδους την παραγωγή. Νομίζω ότι η βιωσιμότητα είναι και θα πρέπει να παραμείνει ο καθοδηγητής όλων των προτάσεων που θέλουμε να ενσωματώσουμε στην έκθεση αυτή. Και βεβαίως εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε και τον ορισμό της βιωσιμότητας, όπως το κάναμε παραδείγματος χάρη με ένα παρόμοιο προϊόν, το κακάο. Και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε και τα τροπικά δάση, αλλά και κάθε άλλους ε, οικότοπους, ε, είτε σημαντικές καλλιέργειες, τις οποίες δεν θέλουμε να καταστρέψουμε. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε καύσιμα, είτε είναι βιοκαύσιμα, είτε κάτι άλλο, πρέπει να αναρωτιόμαστε για τη βιωσιμότητα ε, της παραγωγής τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση για τις 8 Δεκεμβρίου για το κοκτέιλ φυσικά και θα παρευρεθούμε. Έπειτα, μια που πρόκειται για το φινικέλαιο, πρέπει να σας πω ότι η Ολλανδία για το 2020 έχει προβλέψει να έχει μόνο φινικέλαιο από βιώσιμες πηγές. Όντω δεν πρέπει να καταστρέφονται τα τροπικά δάση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά φυσικά και πρέπει να βοηθήσουμε και για τη διατροφή του κόσμου, που σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ε, βούτυρο ή άλλα έλαια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμες παραγωγές αντί για το φινικέλαιο. Αλλά πρέπει να βρούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Και όσον αφορά τώρα τη συνειδητοποίηση για την βιοπικιλότητα, και τα τροπικά δάση στον τρίτο κόσμο και εδώ πρέπει να συνεργαστούμε και να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση που έχουμε κάνει και παλιότερα σε μια άλλη αίθουσα. Δεν θέλω να πω Φυσικά και ούτε μου αρέσει να λέμε ότι είμαστε κατά του φινικέλεου, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και την οικολογία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο και ξανά για τα τροπικά δάση. Ευχαριστούμε, κύριο Σταφρόντε. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Εύη είναι σχεδόν συγκεντρία και ε, μου είπε στη θέση της. Να πω τα εξή πρώτα από τα συγχαρητήρια για την έκθεση στην εισηγήτρια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή το κειμενό τη και συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση. Και επίσης ε, συμφωνούμε ιδίω εκεί που λέω ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε ε, αυτό το φινικέλιο το 2020 ακριβώς όπως θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα βιοκαύσιμα μέχρι τότε επίσης στο Στρασβούργο τοποθετήθηκε σχετικά η κυρία Εύη και είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα κάνουμε για το εμπόριο του φινικελαίου γιατί για το κλίμα και για το περιβάλλον υπάρχουν σημαντικές συνέπειες. Άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάτι το βιώσιμο και γι' αυτό και κατεβάζουμε κάποιες τροπολογίες όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης. Επίση πρέπει να τεθούν κάποιες ε, αυστηρές προϋποθέσεις, αυστηρά κριτήρια, όπως είναι το να ελεγχθεί ε, το, η επίπτωση που υπάρχει στο περιβάλλον από αυτή την παραγωγή. Και αυτά τα συστήματα της πιστοποίησης θα πρέπει να αποτελούν εγγύηση ότι δεν θα υπάρχει ε, βλάβαιο για την βιοπικιλία και δεν θα ζημιώνονται επίση και οι θαγενείς πληθυσμοί. Άρα θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει όσον αφορά και τις γέες που χρησιμοποιούνται για αυτή την καλλιέργεια. Και αυτό να λεφθεί υπόψη για την επιστοποίηση. Θα πρέπει επομένως να αποκαταστήσουμε τις βλάβες που έχουν δημιουργηθεί στους οικολογικούς διαδρόμους. Και στην έκθεση του 2011 είχαμε ξαναπεί ότι χρειάζεται να υπάρξουν εγγύσεις βιωσιμότητας για αυτή την ε, ε, παραγωγή και θα πρέπει όλα αυτά να θωρακιστούν με κάποιο σωστό νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρξει εποπτεία του πώς γίνεται η φύτευση, πώς γίνεται η καλλιέργεια ε, αυτού του προϊόντος. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει σε αυτήν την εκθέση να ληφθεί υπόψη όλο το, το, το, πλέγμα των προβλημάτων και για το περιβάλλον αλλά και για τις επιπτώσεις και αυτού του εμπορίου όσον αφορά την ε, φύση και τη βιοποικιλότητα. Για αυτό και εμείς ε, θα έχουμε κάποιες τροπολογίες για τις μη οικονομικές πτυχές του θέματος. Θα πρέπει να γίνει επίσης υποκατάσταση των ε, δασών εκεί που πρέπει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θέλει άλλο το λόγο από τους συντέλφους, όχι από ό,τι φαίνεται. Και τώρα. Κύριε Σαμανούλ Μάιλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την Να συγχαρώ και την εισηγήτρια και όλους όσους έχουν συνεισφέρει στην ε, εργασία αυτή που αφορά το φιλικέλαιο. Αρχικά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν την αποψήλωση. Είδαμε τον κύριο Ναβάρο, ο οποίος μίλησε για τους ε, στόχους ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως το θέμα της καταπολέμησης της αποψήλωσης και καταστροφής των δασών ενσωματώνονται σε αυτούς τους στόχους της ε, αηφόρου ανάπτυξης. Βεβαίως, κάνουμε πολλά για να στηρίξουμε αυτή τη δράση μέσω του προγράμματος FLECT στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, με τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Σύμβασης για την Βιοπικιλότητα, με το πρόγραμμα Red για την δράση Συνθήκη. και όσον αφορά την παράνομη αποψήλωση η κυρία Μογκερίνη συναντά τους υπουργούς εξωτερικών για τις πρώτες άδειες φλεκτ οι οποίες θα είναι έτοιμες ε, και θα φτάσουν στην Ευρώπη σε λίγες μέρες. Μάλιστα έχουμε και τη δέσμευση του Βιετνάμ για την καταπολέμηση της αποψήλωσης. Προτίθεται και το Βιετνάμ να υπογράψει εταιρική σχέση με την Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε από τη μία την νόμιμη καταστροφή των δασών και από την άλλη θέματα υποδομών, καλλιέργειας, επέκταση των αστικών περιοχών. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα δηλαδή. Η αποψήλωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από όλους μας και από τις χώρες στις οποίες υπάρχουν αυτά τα μεγάλα τροπικά δάση, αλλά και από όλους τους ε, δημόσιους ε, φορείς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εργάζονται και προετοιμάζουν μία μελέτη, εξετάζουν τους τρόπους καταπολέμησης της αποψήλωσης και βεβαίως ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, στην, ίσως στην αρχή του 2017. Ιδιαίτερα για το φινικέλαιο, Ξέρετε ότι η πολιτική μας, ε, ειδικά για το φινικέλεο δεν υπάρχει. Γνωρίζουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ε, εδώ, αλλά και από την κοινή γνώμη. Και γνωρίζουμε ότι το φινικέλεο βεβαίως ε, έχει πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, πολύ σημαντικά κέρδη για τους πληθυσμούς των χωρών αυτών που ζουν χάρη στο φινικέλαιο και στην ε, καλλιέργειά τους και είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι για τα θέματα της αποψήλωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε σε ένα διεθνές επίπεδο, να συνεργαστούμε με όλες τις αγορές κατανάλωσης του φινικέλαιου και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και μία καινούρια έρευνα και θα ήθελα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε γι' αυτό, που αφορά τις ε, περιβαλλοντολογικές συνέπειες της καλλιέργειας του φινικέλεου. Πρόκειται για μια δεύτερη μελέτη, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017 και ελπίζουμε χάρη στην δική σας ε, μέχρι τώρα ε, δουλειά για το θέμα του φινικέλου και των επιπτώσεων θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή δράση και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η τρέχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδους και όλους όσους πήραν το λόγο και αναφέρθηκαν στις γνωμοδοτήσεις που περιμένουμε και στις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους όσους μίλησαν για τροπολογίες που θέλουν να υποβάλουν. Εγώ πραγματικά θα συμπεριλάβω όλες τις προτάσεις σας στο κείμενο. Θεωρώ ότι ε, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα κείμενο που αφορά ένα νέο θέμα για το Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό σε μια έκθεση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. για το πώς θα το παρουσιάσουμε. Βεβαίως δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια θέματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολήσουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις προτάσεις. Το θέμα αυτό δεν θα το εξαντλήσουμε με μία μόνο έκθεση, αλλά σίγουρα ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει πολλή πλευρά. Με μεγάλη χαρά θα συνεχίσω τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεωρώ ότι η παραγωγή φινικέλεου η οποία σε γενικές ποσότητες αυξάνεται, θα πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να εκφράσουμε στην έκθεση αυτή της απόψη μας για το πόσο πολύ θέλουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τον περιορισμό της παραγωγής αυτής, και σε ποιες περιπτώσεις το φινικέλαιο είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε, να το στηρίξουμε και ποιες είναι οι περιπτώσεις που θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να απαγορευτεί. Σκοπός μας δεν είναι να απαγορευτεί το φινικέλαιο σαν ουσία, αλλά να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές που θα κάνουν την καλλιέργειά του, την παραγωγή του βιώσιμη. Και βεβαίως μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι κοινωνικές συνέπειες αυτής της παραγωγής. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες και για τους πληθυσμούς που ζουν από αυτήν την παραγωγή, αλλά βεβαίως να δούμε και τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον και να είμαστε σταθμισμένοι και ισορροπημένοι στη δράση μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I have to remember... Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα λάβει χώρα 9 Μαρτίου του 2017. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων της εξοριστικής βιομηχανίας. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή στον κύριο Χούλιο Γκαρσία Πόρκες και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον εισηγητή και τους σκιώδες μας εισηγητές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που δίνετε στην Επιτροπή την ευκαιρία να σας παρουσιάσει εδώ στην Επιτροπή σας την έκθεσή μας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μια σημαντική νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε μετά από κάποια ατυχήματα. Το ένα στη Νότια Ισπανία και το δεύτερο στη Ρουμανία. Κεντρικός και βασικός στόχος είναι να αποφεύγουμε ή να μειώνουμε όσο γίνεται περισσότερο τον κίνδυνο ατυχημάτων από τα απόβλητα των εξορρυκτικών βιομηχανιών. Τα θέματα της ασφάλειας φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικά στην οδηγία. Τώρα έχουμε και τη διάσταση της κυκλικής οικονομίας που αποκτώ και μεγαλύτερη σημασία. Τα απόβλητα από τις εξορρυκτικές βιομηχανίες το 35% των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανακύκλωση ή αποφυγή των αποβλήτων αυτών είναι ένας στόχος που λαμβάνουμε υπόψη όταν πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας. Επιπλέον, στο πρόγραμμα δράσης της κυκλικής πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται δύο πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τις ε, πρωτεσίλες από την εξοριστική βιομηχανία όταν βρίσκονται στα απόβλητα, πώς θα την ε, πάρουμε πίσω, πώς θα πάρουμε πίσω αυτές τις ε, ουσίες. Πώς θα τις ανακτήσουμε. Και αυτό απαιτεί βέβαια περισσότερη δουλειά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή εδώ βασίζεται βέβαια στις τριτής εκθέσεις που υποβάλλουν οι χώρες μέλη. Όμως, έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες πηγές ενημέρωσης. Για παράδειγμα, τις εκθέσεις σχετικά με τα ατυχήματα που έχουν λάβει η χώρα, αλλά και στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες των εθνικών ε, υπηρεσιών. Όλες οι χώρες μέλη έχουν υποβάλει εκθέσεις. Βέβαια είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα, αυτό το αποδεχόμαστε για όλες. Πάντως βλέπουμε ότι εκθέσεις αυτές μερικές φορές δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Είτε γιατί δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας οι χώρες μέλη, είτε για άλλους λόγους. Το καλό νέο πάντως είναι ότι οι εκθέσεις αυτές δείχνουν ότι γενικώ τα μέτρα έχουν εγκριθεί από τις χώρες μέλη και το επίπεδο συμμόρφωσης είναι αυτό που διαφέρει κάπως. Αλλά παρόλα αυτά και αυτό είναι αρκετά καλό. Όμως υπάρχουν και κενά σε διάφορους τομείς. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο αριθμός των εξοριστικών βιομηχανιών που διαθέτει μια χώρα. Δεύτερον, ο αριθμός των κατηγοριών ε, α ή άλλης που έχουν ε, οι χώρες μέλη. Έπειτα η συμμόρφωση, κατά πόσο δηλαδή τα ατυχήματα που γίνονται αναφέρονται πάντα. Για το θέμα των διευκολύνσεων που υπάρχουν για τα απόβλητα, κάποιες εκθέσεις αναφέρουν πολύ χαμηλό αριθμό τέτοιων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Έξι χώρες μέλη λένε ότι δεν έχουν καθόλου τέτοιες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων εξοριστικών ε, βιομηχανιών ε, στην επικράτειά τους. Άλλες όμως πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι αυτές οι χώρες έχουν εξορυκτικές ε, δραστηριότητες που δημιουργούν απόβλητα. Όταν πρόκειται για την κατηγορία Α, εδώ το θέμα της συμμόρφωσης διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Κανονικά υπάρχει υποχρέωση από την οδηγία στην διαφοροποίηση των αποβλήτων, ανάλογα με το πόσο επικίνδυνα είναι, και επιβάλλονται φυσικά πιο αυστηρές ε, προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με απόβλητα υψηλότερου κινδύνου. Σημαντικός αριθμός χωρών ανέφερε ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις κατηγορίας Α στην επικράτειά τους. Όμως, συγχρόνως, κάποιες από τις χώρες αυτές ανέφεραν μεγάλους όγκους επικίνδυνων εξορρυκτικών αποβλήτων. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που δίνουν στις εκθέσεις τους οι χώρες μέλη δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες εφόσον το, η επικινδυνότητα των αποβλήτων αυτών είναι απόδειξη για την ύπαρξη κατηγορίας Α. Επιπλέον το 25% των εγκαταστάσεων ε, κατηγορίας Α ε, δεν έχουν πάντα συστήματα ε, διοχέτευσης των αποβλήτων αυτών. Έπειτα υπάρχει το θέμα των αδειών στην οδηγία που συνδέεται μερικές φορές με τις απαιτήσεις για πιστοποίηση άλλων οδηγιών, σοβέζο για παράδειγμα. Οι εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται στην, ε, σε εκθέσεις αυτές είναι συχνά κατηγορία σοβέζο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται περισσότερη έρευνα και διευκρίνηση. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις τώρα, οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών βιομηχανιών υποχρεωτικά πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ακόμα και αφού έχει κλείσει η εγκατάσταση. Η έκθεση όμως δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών μελών και από αυτού όσον αφορά τη φύση των επιθεωρήσεων, όσον αφορά τη συχνότητα των επιθεωρήσεων και επιπλέον κάποιες χώρες μέλη ανέφεραν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους της άδεια την περίοδο 2011 με 2014. Είναι πολύ χαμηλός ε, ο αριθμός, μεν, αλλά μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που δεν εντοπίζονται εξαιτίας της έλλειψης ικανοποιητικών επιθεωρήσεων. Και αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί παρετέρω διερεύνηση. Όσον αφορά τώρα τα ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει περιπτώσεις ατυχημάτων σε τέτοιες εγκαταστάσεις εξορρυκτικής βιομηχανίας, όμως τα ατυχήματα αυτά δεν αναφέρονται πάντα στις αιτήσει κοινοποίησης βάσει υποχρέωσης που έχουν οι χώρες μέλη. Οπότε τις πληροφορίες αυτές χρειάστηκε να τις πάρουμε από τα μέσα ενημέρωσης ή από άλλους φορείς. Εν κατακλείδη, θα έλεγα, Πρόεδρε, ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα πόβλητα από την εξωτική βιομηχανία, παραμένουν όμως ελλείψεις. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι στόχοι της οδηγίας να υλοποιηθούν. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει, που θα αρχίσουν σύντομα. Πρώτον, ενημερώνουμε το έγγραφο αναφοράς όσον αφορά τι βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές όσον αφορά τα απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας. Η διαδικασία άρχισε πριν από δύο χρόνια ήδη και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά. Δεύτερον, φέτος αρχίσαμε μια πρωτοβουλία πρόθεσης της συμμόρφωσης προκειμένου να εντοπίσουμε τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και προκειμένου επίσης να εντοπίσουμε βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή που στη συνέχεια βέβαια ε, τις δίνουμε και στις υπόλοιπες χώρες μέλη. Επίσης θέλουμε να καταγραφούν όλες οι εγκαταστάσεις. Είναι και αυτή μια δυνατότητα πάνω στην οποία προβληματιζόμαστε. Τρίτον, σε συνεργασία με του εμπειρογνώμονε των χωρών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντοπίσει ζητήματα ή τομείς όπου η τομεί οπου η ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Και στη συνέχεια θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές το 2018. Επίσης το 2018 θα ετοιμάσουμε κατευθυντήριες γραμμές και για επιθεωρήσεις σε συνεργασία κατά πάσα πιθανότητα με το δίκτυο επιθεωρητών για το περιβάλλον. Αυτά πρόεδρε, αλλά ίσως πριν ολοκληρώσω να σας πω ότι εντοπίσαμε ένα μικρό λάθος στην έκθεσή μας. Υπάρχει η κατηγορία Α και σχετικές εγκαταστάσεις, η Πολωνία μας ενημέρωσε για αυτές, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στην έκθεσή μας. Σύντομα θα υπάρξει διορθωτικό. Αυτά είναι όλα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε εισηγητές και σιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να σας το πω στα ουγγρικά, τη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Χόλβενη, και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώ απαντώντας καταφατικά. Είναι αλήθεια ότι επί πολύ περιμέναμε για να αναλύσουμε αυτήν την οδηγία Μπράβο για τη δουλειά που κάνατε γιατί απέτησε πολύ κόπο. Και να σας ευχαριστήσουμε και για την συνεργασία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία για τα απόβλητα της εξορρυκτικής βιομηχανίας με λύσαν προσεκτικά, τον με το έγγραφο και τον καταλαβαίνουμε γιατί μα πήρε τόσο χρόνο να, να, να, επιληφθούμε, γιατί δεν ήταν εύκολο. Με τίποτε θα ήθελα να είμαι στη θέση σα. Και κυρίω. Ξέρω ότι σε μία τριετία δύο φορές κάνατε την ίδια δουλειά. Γιατί τα κράτη-μέλη εξέδεσαν την οδηγία, μετά πήγαν να την εφαρμόσουν, αλλά ο καθένας έκανε το κεφαλιού του, οπότε δεν ήταν εύκολο έτσι να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα του τοπίου για την εφαρμογή και τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, οπότε όπως και σε άλλες οδηγίες καταλήγουμε στο ίδιο. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να βλέπει στην πράξη που καταλήγει κάθε οδηγία. Ποτέ λοιπόν μας κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει με το που θεσπίζεται ένα νομοθέτημα. Θα πρέπει να περιμένει την ώρα της εφαρμογής. Το 2006 λέει θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα έχουμε ε, την, την ανάλυση κάποιων αρνητικών συνεπειών όσον αφορά το τοπίο, τη φύση, ε, την πανίδα, τη χλωρίδα για να αναλύσουμε ποιοι είναι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και έτσι να δούμε τι θα γίνει με την ε, διαχείριση ε, αυτών των αποβλήτων της εξωτερικής βιομηχανίας. Οπότε, τελικά το θέμα δεν είναι το κατά πόσον κάποια κρατημέλη θα εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους, πώς θα γίνεται η ενημέρωση των εμπλεκομένων. Το θέμα είναι άλλο. Είναι το εξή. Αν θα μπορούσαμε να ζούμε μέσα σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. στο θεματολόγιο του Κοινοβουλίου ανέκαθεν ήταν το θέμα των επιπτώσεων τη εκκροτικής βιομηχανία πάντω, ανέκαθεν ε, από πλευρά δική μα το ερώτημα, είναι ασφαλή η Ευρωπαία από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του είδου τη τεχνολογία και ιδίω όσον αφορά τα απόβλητα. Και για να διασκεδαστούν αυτέ οι ανησυχίε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα λέει τα ίδια. Δηλαδή, ότι η οδηγία εξασφαλίζει την, ε, το, το να μην υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει από αυτέ τι δραστηριότητε και ότι είναι επαρκή η σχετική νομοθεσία. Εάν εφαρμοστεί όπω πρέπει και έτσι δεν θα έχουμε ατυχήματα και τι αντίστοιχε συνέπειε αυτών. Άρα, κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα. Και δηλαδή να δούμε ακριβώ πού δεν τα πήγε καλά η εφαρμογή, να δούμε κατά πόσον αυτή η οδηγία καταφέρνει φέρνει το σκοπό της. Στην έκθεσή μου θα σας τα αναλύσω. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αναλυθούν πληροφορίες των κρατών Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητε του σήμερα, του σήμερα ισχυόντος συστήματος της αναφοράς προς την ε, Επιτροπή. Άρα όλα αυτά τα μέτρα θα δοκιμάσουν στην πράξη. Επίσης και τα άλλα γενικά μέτρα για να υλοποιηθεί αυτή η οδηγία. Αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν προσαρμοστεί και ενταχθεί στο δίκαιο των περισσότερων κρατών μελών. Οπότε και η εφαρμογή αλλά και η ερμηνεία των σχετικών ορισμών και των διατάξεων που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και έτσι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι και πολύ αξιόπιστα. Αυτά για την οδηγία όλα. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εκεί δεν καθορίζεται το πώς θα γίνονται. Οπότε, αποτελεί κοινό μυστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιε κατευθύνες γραμμές για αυτές τις επιθεωρήσει. Έχουμε το άρθρο 22 το οποίο η έκθεση ορθώς το αναφέρει και αυτές οι κατευθυντήριε σίγουρα βελτιώνουν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των σχετικών εγκαταστάσεων για όλα τα κράτη-μέλη. Πέραν όλων αυτών τώρα που είναι πολύ σημαντικά, με δύο λόγια να σας τονίσω κάποια άλλα σημεία τα οποία και στην έκθεσή μου θα τα αναπτύξω και αυτά. Αυτά τα απόβλητα από την εξωτερική βιομηχανία αποτελούν το 30% των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν, τι προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με αυτόν τον οικονομικό κύκλο. Και να δούμε τι εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν, τι τεχνολογίες υπάρχουν για το περιβάλλον και έτσι να μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των απόβλητων της εξωτερική δραστηριότητας. Και δεν μιλάμε βέβαια για κατάργηση αυτής της δραστηριότητας. Ξέρουμε όλοι το πόσο χρειάζεται και τόσο χρειάζονται τα προϊόντα αυτής. Χρειάζεται όμως να γίνει σωστή εφαρμογή των κανόνων με τρόπο αυστηρό. Τελευταίο αλλά σημαντικό. Συνήθως όταν έχουμε την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων υπάρχουν δεσμένες συνέπειες για τις ντόπιε κοινότητες και τον κόσμο που ζει εκεί. Οπότε και τόσα χρόνια έχουμε προσπαθήσει κάτι να κάνουμε με τις ε, εφαρμοστικές εκθέσεις. Συνεχίζω στα ουγγρικά τώρα. Συνάδελφοι, πολλά είναι τα ερωτήματα που μένουν απάντητα. Τώρα δεν έχουμε τον χρόνο να τα θίξουμε όλα. Όμως είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στο γραφείο μου να έρθετε να με βρείτε γιατί περιμένω πώς και πώς τις παρατηρήσεις σας ε, και εγώ και οι συνεργάτες μου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση με την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Έχουμε επίσης και την ε, υπηρεσία έρευνα στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι μας βοηθούν με πολύ υλικό έρευνας και έτσι θα συνεχίσουμε τις επαφές με τους συναδέλφους τέλο πάντων με την, με την βιομηχανία αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τη γνώμη όσο γίνεται περισσότερων. Άρα, θα προσέξουμε τι θα γίνει με την προσέγγιση του περιβάλλοντος, θα γίνει με την ασφάλεια και πώς θα έχουμε και αποτελεσματικότητα ε, στο σχετικό κλάδο της βιομηχανίας. Και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κονέτσινα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και όλους τους συναδέλφους. Αναφέρθηκαν κάποια πράγματα που κι εγώ ήθελα να πω. Θα συμπληρώσω απλώς με δύο σημεία. Πρώτον, το θέμα των οικονομικών εγγύσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά ή αρκετά υψηλές έτσι ώστε να καλύψουν όλα τα πιθανά, αν θέλετε, ε, όλες τις πιθανές ε, βλάβες από μια τέτοια εξορρυκτική δραστηριότητα. Πιστεύω δηλαδή ότι τα ατυχήματα που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες μας δείχνουν ότι θα πρέπει σίγουρα να είμαστε πιο προσεκτικοί και να δώσουμε πολύ περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια. Ξέρουμε ότι οι τραγωδίες αυτές κοστίζουν όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές, αλλά πλήττουν και το περιβάλλον. Και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι ορολογιακές βόμβες οι οποίες αργά ή γρήγορα μπορεί να οδηγήσουν σε τραγωδίες, σε θύματα και σε καταστροφές του περιβάλλοντος. Ίσως λοιπόν αυτά που γνωρίζουμε σήμερα να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη χρήση των αποζημιώσεων. Αλλά, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, το θέμα της πρόληψης, το θέμα των επιθεωρήσεων του ελέγχου που γίνεται επιτόπου και της παρακολούθησης. Αυτό θα πρέπει να γίνεται και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά από και εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται βάσει πολύ συγκεκριμένων εργαλείων και κριτηρίων συγκρίσιμων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να εντατικοποιηθεί στο μέλλον έτσι ώστε όταν μιλάμε για απόβλητα να χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές τεχνολογίες έτσι ώστε να γίνεται η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων και εκεί όπου αυτό είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιούνται σε κυκλώματα παραγωγής. Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της δραστηριότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Ντορνανό. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να δώσουμε ιδιαίτερη προσφυγή σε αυτά τα απόβλητα που απορρέουν από την ε, εξορρυκτική δραστηριότητα. Είναι περίπου το 30% των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να αποφύγουμε τη μόλυνση και να αποφύγουμε και τα ατυχήματα. Η οδηγία του 2006 μα έδειξε ότι τα 10 τελευταία χρόνια υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίε και αδυναμίες όσον αφορά την ε, μεταφορά του κειμένου τη οδηγία στην Ομοθεσία των κρατών μελών. 22 αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες και πολλές προσφυγές για την μη συμμόρφωση έχουν αναφερθεί μέσα σε αυτήν την δεκαετία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές χώρες όπως η Λετωνία, η Λιθουανία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ολλανδία δεν έχουν εγκαταστάσεις που να μπορούν να συμμορφωθούν με αυτές τις προδιαγραφές. Βλέπουμε λοιπόν ότι άλλες πηγές αναφέρουν το αντίθετο, υπάρχει λοιπόν μεγάλη σύγχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ε, ομοιόμορφη και ενιαία εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αυτό όμως είναι αντίθετο με το πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών. Όπως ξέρετε θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην κάθε οδηγία και να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα της επιλογής τους, τα εργαλεία της επιλογής τους για την υλοποίησή της. Αντί λοιπόν να απορούμε γιατί υπάρχουν διαφορετικοί ε, μέθοδοι, διαφορετικά στοιχεία, διαφορετική επεξεργασία τελικά των αποβλήτων, ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε και να αμφισβητήσουμε τη μέθοδό μας, γιατί εδώ πρόκειται για μια απλή οδηγία, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και πολύ περιοριστική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να σεβαστούμε περισσότερο τις επιθυμίες και τα αποτελέσματα των κρατών μελών, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ έξω για να μιλήσω εξ ονόματος της σκιώδους εισηγήτριας, η οποία δεν είναι παρούσα, και να μιλήσω για την χρήση των αποβλήτων στην κυκλική οικονομία. Από την αρχή της συζήτησής μας για την αναθεώρηση του κειμένου της οδηγίας, θεωρήσαμε ότι η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν στην κυκλική οικονομία όλα αυτά τα απόβλητα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Συνεχίζω. Δεν θα ξαναρχίσω την αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία του 2006 21, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα απόβλητα και την επεξεργασία τους, απόβλητα που προέρχονται από την εξορρυκτική δραστηριότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία από τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη αναφορά και πολύ πιο ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας. Προτείνει μια λύση ουσιαστικά η Επιτροπή με τις κατευθυντήριες γραμμές και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να υιοθετήσουμε σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Το άρθρο 5 της οδηγίας που αφορά με σχέδια επεξεργασίας αποβλήτων αναφέρεται στη μείωση των αποβλήτων, στην πρόληψη, καθώς και στην ανακύκλωση από την άλλη. Η Επιτροπή έχει συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το θέμα της πρόληψης και της ανακύκλωσης χρησιμοποίησης των αποβλήπεων. Πώς δηλαδή έχουν τα πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Να ξαναδώσουμε λοιπόν το λόγο στην Επιτροπή για να δώσει μια απάντηση και να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν άκουσα ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός μία. Συμφωνώ πάντως με τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας η κυκλική οικονομία, η διάσταση της κυκλικής οικονομίας σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είπα, έχουμε δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αυτό το οποίο προβλέπετε σε αυτήν την ε, ε, προσπάθεια του προγράμματος δράσης για την κυκλική οικονομία και η οδηγία για αυτού τους καταστροφικά απόβλητα εκεί εστιάζει την προσοχή της αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ε, παραβλέψουμε τις ε, απόψεις του θέματος που έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία γιατί και εκεί τα πράγματα έχουν μεγάλη σημασία τώρα όσον αφορά την ε, χρησιμότητα αυτού του μηχανισμού που προβλέπει η οδηγία ξέρετε η εμπειρία μας από τους μηχανισμούς υποβολής ε, εκθέσεων δεν είναι κάτι το τόσο ενθαρρυντικό. Στη σχετική μας πρόταση είχαμε πει ότι θα πρέπει να απαλληφθούν κάποιες ε, προϋποθέσεις και κάποιες ε, ε, οδηγίες όπως η οδηγία για τις χωματερές, η οδηγία για τη συσκευασία ε, αλλά η συγκεκριμένη οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική και χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ε, υποβολής των εκθέσεων. Α, πρέπει να αναφέρονται τα ατυχήματα. Το θέμα επίσης των χρηματικών εγγύσεων έχει τεθεί. Και σήμερα με την οδηγία προβλέπεται τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν τέτοια συστήματα χρηματικών εγγύσεων. Δυστυχώ, αυτή η δυνατότητα δεν έχει αξιοποιηθεί. Τώρα, όσον αφορά τη μεταφορά τη οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, ξέρετε ότι αυτό ήταν ένα από τα δύσκολα σημεία ξεκίνησαμε διαδικασία παραβάση για 25 ε, ε, ε, διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν έγινε, δεν ολοκληρώθηκε σχετική διαδικασία. Αυτά μέχρι το 2011. Αλλά λίγα χρόνια μετά από την κατακλητική ημερομηνία όπως οριζόταν στην οδηγία. Πάντως, Δεν νομίζω ότι τέτοιοι μηχανισμοί και οικονομικά κίνητρα θα είναι τόσο αποτελεσματικά όσο το να υπάρχει ένα σωστό αυθεντικό κανονιστικό πλαίσιο. Και όσο αφορά την ασφαλεία των εγκαταστάσεων. Τώρα, μα επιθύνεται κάποια ερώτηση όσον το άρθρο 5 και τη διαχείριση των αποβλήτων και την προληπτική δράση. Ναι, όντω αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση για το πώς αυτό έχει ληφθεί υπόψη στα προγράμματα διαχείρισης ε, των αποβλήτων ακριβώς για αυτό και ε, το έχουμε αυτό για την πρωτοβουλία μας ως βασικό στόχο. Η αλήθεια είναι πως ότι κάτι ήδη έχουμε ξεκινήσει σαν πρωτοβουλία και τον Μάρτιο του χρόνου θα γίνει το πρώτο εργαστήρι όπου θα συμμετάσχουν τα κρατημέλη και οι εμπλεκόμενοι. Τέλο πάντων, αυτό είναι το τελευταίο που έχω να σα πω και με μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με, την, με τον εισηγητή, γιατί έχει μπροστά του δύσκολο έργο. Μπορεί να υπολογίζει σε εμάς. Ε, ευχαριστώ. Ε, εγώ λέω ο Οπότε εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε τη για αυτό το σημείο στην ημέρα και μπορούμε να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα το οποίο είναι η ανταλλαγή απόψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ΣΥΤΑ. Η κυρία Μπάσκα θα μας τα πει από πλευρά τη ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπάσκα είναι η επικεφαλή διαπραγματεύτρια για τη συνθήκη με τον Καναδά. Yes. For starting Θα uh, αρχίσουμε τη συζήτηση με την ε, εισήγησή σας και στη συνέχεια να ακούσουμε και έχουν πει, να πούν οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, πώς βλέπουμε τα πράγματα σε σχέση με τη ΣΥΤΑ και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και κάποιες ε, ερωτήσεις. Σύντομα λοιπόν να σας πω ότι θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά την αύξηση των ευκαιριών για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις και αυτό σαν αποτέλεσμα των ε, προσπαθειών μας να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη. Είναι η πιο προοδευτική επίσης συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί και υπογράψει όσον αφορά την πρόσβαση στις αγοράς, στις αγορές, συγγνώμη, σε αυτή τη συμφωνία από την πρώτη κιόλας ημέρα οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες με τη μείωση των δασμών, με την προστασία των πιο ευαίσθητων κατηγοριών γεωργικών προϊόντων, με ειδικέ ε, δεσμεύσεις για κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα και κατηγορίες που θα εισάγονται. Τώρα, ανοίγει όχι μόνο η αγορά των ε, υπηρεσιών, αλλά και κάποιοι άλλοι παράγοντες και τομείς όπως ε, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι προμήθειες, παραδείγματος χάρη στον Καναδά, είναι ένας από τους τομείς που ανοίγουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες νέες δυνατότητες. Η συμφωνία αυτή διατηρεί και προστατεύει τις ε, θεμελιώδες αξίες για μας, όπως φόρος ανάπτυξη, βιωσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για αξίες οι οποίες εμπεριέχονται σε αυτή τη νέα συμφωνία και βεβαίως πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία με δεσμευτικές και όσον αφορά την εργασία βασιστήκαμε στα κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και ο προοδευτικός χαρακτήρας αυτής της συμφωνίας ε, ενισχύεται από την ε, ενσωμάτωση ε, συμφωνία, στη συμφωνία αυτή διατάξεων για τις επιχειρήσεις, για την επίλυση των διαφορών, τα μηνύματα που δεχόμαστε σήμερα από τον Καναδά είναι ότι συμφωνεί και συμμορφώνεται και εναρμονίζεται πλήρως με την στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στα πλαίσια της πολυμερούς αυτής συμφωνίας θέλουμε να βελτιώσουμε το συνολικό σύστημα επίλυσης διαφορών σε θέματα επιχειρησιακά και επενδύσεων, όχι μόνο δηλαδή με τον Καναδά, αλλά και διεθνώς. Το τελευταίο στοιχείο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τον προοδευτικό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας, είναι το γεγονός ότι τα δύο συμβαλόμενα μέρη προστατεύουν το δικαίωμα του καθορισμού, της προστασίας, κάποιων δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων στον δημόσιο τομέα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά ο δημόσιος τομέας, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ίστατο αγαθό. Ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα η διαδικασία της κύρωσης είναι μια δύσκολη, περίπλοκη διαδικασία, χρονοβόρα και με μεγάλη χαρά ε, θα απαντήσω τυχόν ερωτήσεις μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής εδώ στο Κοινοβούλιο. Αν χρειάζεσαι κάποιες διευκρινήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζουμε ότι η ανταπόκριση του Κοινοβουλίου θα είναι ταχύτατη και ότι το συντομότερο δυνατόν θα μπορέσουμε να εποφαληθούμε ε, εμείς και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τα θετικά αυτής της συμφωνίας. Όσον αφορά την διαδικασία κύρωσης, σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν ε, ερωτηματικά που αφορούν κυρίως το δημόσιο τομέα, την προστασία των επενδύσεων. Πραγματικά ηγετικό ρόλο εδώ έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς συμφώνησε, συμμορφώθηκε, πρόκειται επαναλαμβάνω για μια φιλολόδοξη προοδευτική συμφωνία συμφωνήσαμε, όπως ξέρετε, και στο διμερές εργαλείο, το οποίο θετήθηκε ε, στην ε, Σύνοδο Κορυφής, στη Διμερή Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Πρόκειται για το υψηλού επίπεδου ε, ερμηνευτικό εργαλείο της συμφωνίας, κάτι που δέχτηκαν και οι δύο πλευρές. Ευχαριστούμε. Το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Στάις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Βασκάρτη, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας και για όσα μας είπατε για την ε, ΣΕΤΑ, που σίγουρα δεν είναι λέτε ότι είναι η πιο σύγχρονη, μάλλον πιο προοδευτική συμφωνία που είχαμε ποτέ, ότι λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα, ότι έχει, αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις βάσει συμφωνιών σε διεθνές επίπεδο. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό. Ένα παράδειγμα είναι το κόντεξ αλιμεντάριους. Όλοι ξέρουμε ότι για τα παρασιτοκτόνα, για παράδειγμα, ο κώδικας αυτός έχει πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές από τις προδιαγραφές που έχουμε εμεί τους δικού μας κανονισμούς που έχουμε γκρίνει το 2009 και άλλοτε. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, μια άποψη για το πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, πώς θα έχουμε τις διάφορες προδιαγραφές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μερικές φορές παρουσιάζει το, τη συμφωνία αυτή έτα σαν να είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ε, κυρωθεί, συμφωνηθεί και έχει τελειώσει. Δεν είναι όμω έτσι. Η συζήτηση, για παράδειγμα, για τους γενετικά τροπομένους οργανισμούς. Ο Καναδάς φυσικά είναι μια χώρα η οποία θέλει την τεχνολογία αυτή και παράγει τέτοια προϊόντα σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι σε αντίθεση με αυτό που θέλουν οι πολίτες και σε αντίθεση με την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των χωρών μελών, ε, λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πίεση τέτοιων ε, εμπορικών ε, συμφωνιών με τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ενόψη μάλλον τέτοιων συμφωνιών, πιέζει για να επιτραπεί η χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα και την επιτρέψει την εισαγωγή τους ε, στην Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε τι έγινε και με τα καύσιμα. Ξέρουμε το ιστορικό. Και τότε υπήρξε πίεση από τον Καναδά για να εξάγουν ε, ε, τέτοια καύσιμα που είναι... αυτήν την άμμο με πίσα. Και θέλω να πω με αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά υποχωρεί για πράγματα όπως τότε τα καύσιμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συζήτηση που είχαμε για τοξικές ε, ουσίες που προκαλούν ε, καρκίνο. Μιλήσαμε επίσης για τους ορμονικούς διαταράκτες. Πάλι υπήρξε διάσταση ανάμεσα στον Καναδά και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Αύριο θα μιλήσουμε για τους ορμονικούς διαταράκτες, ε, Πρόεδρε. Διότι φαίνεται να προχωρούν τα πράγματα όπως θέλει ο Καναδάς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά από την πίσω πόρτα βάζει πράγματα τα οποία εμείς και η δικιά μας νομική υπηρεσία ε, βρίσκει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Και κάτι άλλο επηρεάζεται η νομοθεσία μας, οι προδιαγραφές μας. Το ΣΕΤΑ δεν έχει υπογραφεί. Τι θα συμβεί λοιπόν άμα αρχίσει να ισχύει η ΣΕΤΑ. Δεν θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ο πρώτος στόχος είναι να μειωθούν οι εμπορικές προδιαγραφές. Μα πώς θα γίνει, τη στιγμή που έχουμε προδιαγραφές, έχουμε στάνταρτ, έχουμε νόμους, για την ασφάλεια τροφίμων, για παράδειγμα. Ε, λοιπόν, πολλοί από αυτούς τους κανόνες είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι είναι για τον Καναδά. Τι θα κάνουμε, τις δικέ μας τι προδιαγραφές ε, θα μειώσουμε και θα καταργήσουμε. Η Συμφωνία ΣΕΤΑ προβλέπει συνεργασία σε θελοντική βάση και δεν υπάρχει υποχρέωση όπως θέλουμε εμείς για τη συμμόρφωση. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία ήδη συμβαίνουν ενώ δεν έχει υπογραφεί καν ακόμα η συμφωνία πλήρως. Και ο μηχανισμός ε, στον οποίο αναφερθήκατε, διαιτησίας, εντάξει, το είπατε, είναι βέβαια μια βελτίωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μηχανισμό διατησίας που είχαμε σε προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, εντάξει, συμφωνώ, όμως τελικά παραμένει να ευνοεί τους επενδυτές και τους δίνει δικαιώματα που άλλοι δεν έχουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γράφονται στη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Τελικά δηλαδή θα είναι οι επενδυτές οι οποίοι θα μπορούν να προσφύγουν σε βάρος χωρών για την ομοθεσία τους. Πέρα από όλα αυτά, Έχω τρεις ερωτήσεις ως εισηγητής προς εσάς, κυρία μου. Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε τα προνόμια μας να διατηρηθούν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνομοθέτης. Το άρθρο 218 της Εθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα πλήρως πρέπει να ενημερώνεται σε όλα τα στάδια τέτοιων διεθνών συμφωνιών και ότι για ευαίσθητα ζητήματα διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται. Τον Απρίλιο υπήρξε μία διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για καλύτερη νομοθέτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή πρέπει πλήρως να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε τέτοιες συμφωνίες. Λοιπόν, σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα κυρία Βασκάρ. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα υπάρξει εγγύηση ότι θα γίνει αυτό πριν υπογραφεί το ΣΕΤΑ, δηλαδή ότι θα τηρηθεί το άρθρο 218.10 που λέει ότι πρέπει πάντα να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ό,τι συμβαίνει στη ΣΕΤΑ. Δεύτερον, διαβάζω στο έγγραφο της ΣΕΤΑ, στο άρθρο 23, ότι υπάρχει, δημιουργήθηκε μια κοινή επιτροπή η οποία μπορεί να πάρει αποφάσεις δεσμευτικές νομικά, μπορεί δηλαδή να αποφασίσει για πράγματα τα οποία θα υπερισχύουν, γιατί θα είναι διεθνής νομοθεσία, θα υπερισχύουν του ε, παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει αυτό. Και τρίτον, μπορείτε να μας εγγυθείτε ότι κάθε φορά που θα τίθεται θέμα προσαρμογής νομοθεσίας θα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν πάρει αποφάσεις αυτή η μεικτή επιτροπή, αυτή η Joint Committee. Δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σαν παγοθράφστη. Δεν πρέπει αυτή να φροντίζει να αλλάζει νομοθεσία χωρίς προηγουμένως να έχουμε συμφωνήσει εμείς. Και τέλος, το άρθρο 30 της ΕΤΑ λέει ότι η μεικτή αυτή η επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει παραρτήματα και πρωτόκολλα. Όχι όλα, αλλά κάποια. Για παράδειγμα, εκείνο που έχει να κάνει με τα φυτογενομικά μέτρα είναι ένα από αυτά. Για μας αυτό είναι βασικό στοιχείο της νομοθεσίας μας και για τη δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Οπότε σας ρωτάω, πώς θα ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πάντα και να μπορεί να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τροποποίησης παραρτημάτων και πρωτοκόλων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά για το δικό μας νομοθετικό έργο εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ωραία. Τώρα θα αρχίσουμε το συνήθι γύρω ομιλητών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Γκάμπους πρώτα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν με τι άλλο πιστεύω ότι είναι καλό να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Είπαμε ότι γίνεται ένας αγώνας κατά του χρόνου, ότι θέλουμε να τελειώσουν ή θέλαμε μάλλον να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις πριν από δύο χρόνια, όμως εμείς τον Ιούνιο πήραμε το πακέτο το νομοθετικό αυτό. Και υπάρχουν και άλλες επιτροπές, η ΙΝΤΑ που επίσης πρέπει να αποφανθεί, καθώς επίσης και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος τέσσερα χρόνια, ε, τέσσερις μήνες αργότερα από τις άλλες επιτροπές εκδήλωσε ενδιαφέρον, δύο εβδομάδες πριν την υπογραφή στο Συμβούλιο. Υπόθηκε ότι θα ιδιωτικοποιηθούν οι πόροι. Στη σελίδα 3 λέει ότι οι διατάξεις δίνουν το δικαίωμα στα διάφορα μέρη να ρυθμίσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα, πολιτισμό κτλ. Επίσης ότι στόχος είναι η προστασία των επενδύσεων των επενδυτών ώστε να μπορούν να κάνουν επενδύσεις, να υπάρξει πρόθεση επίσης της κοινωνικής ευθύνης στη δικαιοδοσία τους. Αναφέρεται η ιδιωτικοποίηση του ύδατος, ενώ το άρθρο 1 λέει ότι δεν είναι ούτε αγαθό ούτε προϊόν. Ότι είναι ένας φυσικός πόρος, το ίδιο ισχύει για τις λίμνες δεξαμενές, όλα τα υδρογραφικά στοιχεία, δεν είναι ούτε αγαθό ούτε προϊόν. Και τίποτα στη συμφωνία αυτή δεν υποχρώνει καμία πλευρά να επιβάλλει την εμπορική χρήση του ύδατος. Πολλά τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να δώσουμε στη συζήτηση αυτή. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε με ναι ή όχι. Οι διάφορες συζητήσεις έχουν ήδη γίνει. Για την ομάδα μας, και δεν θα επεκταθώ πολύ, πρέπει να αποφασίσουμε ναι ή όχι και όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε τώρα το χρόνο να κάνουμε άλλου είδους συζητήσεις. Ο χρόνος αυτός έχει περάσει, έχει παρέλθει. Η θέση μας είναι σαφής και είναι υπέρ αυτής της εμπορικής συμφωνίας. Ευχαριστώ. εκ μέρους των σοσιαλιστών. Τώρα κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις και να μας δώσει απαντήσεις. Σίγουρα χρειάζεται έλεγχος της εμπορικής συμφωνίας και να βρεθεί ένα συμβασμός και η διαφάνεια επίση είναι ζωτική συμφωνία, όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, αλλά για οποιαδήποτε συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι εμπορικέ συμφωνίε στηρούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προστατεύουν το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα για τα οποία είμαστε εμεί υπεύθυνοι στην Επιτροπή μα εδώ. Και θα αρχίσω με τις διατάξεις για το περιβάλλον της ΕΤΑ. Γιατί αυτές λένε ότι τα διάφορα μέρη πρέπει να φροντίζουν για τα επίπεδα προστασίας. Αν λοιπόν αποτελέσει μοντέλο πρότυπο για τις εμπορικές ε, συμφωνίες η ΣΕΤΑ, γιατί δεν περιλαμβάνει τις προδιαγραφές ε, άλλων εμπορικών συμφωνιών όσον αφορά το περιβάλλον. Για παράδειγμα, εξάγει πετρέλαιο ο Καναδάς ε, με τη μορφή της ε, άμμου πίσας, κάτι το οποίο για μας έχει μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θέλω λοιπόν να ξέρω, η ΣΕΤΑ θα αποθαρρύνει τέτοιου είδους πηγές που καταστρέφουν το περιβάλλον και τι ρήτρες ασφαλείας υπάρχουν από αυτού. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει την διευθέτηση ε, διαφωνιών με το νέο σύστημα διατησίας. Για το περιβάλλον όμως δεν υπάρχει αντίστοιχος μηχανισμός διατησίας. Πώς βλέπει ρεαλιστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό της διευθέτησης διαφωνιών όταν πρόκειται για το περιβάλλον. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με την προσέγγιση όσον αφορά τα τρόφιμα για την ασφάλεια τροφίμων. Και το ρωτάω γιατί ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετική προσέγγιση για τη σχετική νομοθεσία. Κυρίως για τις άδειες, τις πιστοποίησεις δηλαδή, τις ετικέτες και τους ελέγχους που γίνονται και το κατά πόσο υπάρχουν ή όχι γενικά δομημένοι οργανισμοί, για την ε, χνηλάτιση του κρέατος, για τα κλωνοποιημένα προϊόντα κτλ. Εδώ υπονομεύεται η αρχή της προφύλαξης, όπως επίσης και η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αγρό στο τραπέζι μας. Πώς θα διασφαλιστούν αυτές οι αρχές στη ΣΕΤΑ. Τέλος. Το δικαίωμα της Μικτής Επιτροπής να εγκρίνει ερμηνεία ή τροποποίηση σε κάποια παραρτήματα και πρωτόκολλα της ε, ΣΕΤΑ χωρίς την ε, δικιά μας παρέμβαση, τα φυτογενομικά μέτρα δηλαδή και τα λοιπά. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς περιμένουν ότι θα αντιδράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για τις Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Αγγέλη, για την Ισία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας πω και πολλά για το θέμα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά τα ακούσαμε και ε, πάρα πολύ καλή αρχή έγινε από τον εισηγητή και έχουμε γίνει το σημείο που μας δίδει στην περσμένη εβδομάδα και τα ακούσαμε και σήμερα το απόγευμα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο μέχρι το αύριο αποφασιστεί τι διαδικασία θα ακολουθηθεί ούτως ώστε να γνωμοδοτήσουμε για μην είναι μαύρο άσπρο. Ναι, όχι. τόσο πάντων να μην χάνουμε το χρόνο μας πάντω από δική μας πλευρά, Είμαι θα υπέρ τη συμφωνία με τον Καναδά και αναγνωρίζουμε ότι έχει καταβληθεί πολύ κόπος για να φτάσουμε εκεί και επίσης ε, ε, άλλοι με, συνέπεια και συνέχεια προσπαθούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία και από το Κοινοβούλιο αλλά και από αλλού. Οπότε τελικά φτάνουμε στο σημείο που θα πρέπει να κλειστεί συμφωνία. Ιδάλλως νομίζω ότι η φήμη μας, ό του Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την σύναψη τέτοιων συνθήκων, πρόκειται να μαυρωθεί πάρα πολύ, γιατί ήδη, ήδη ε, παραπέρασε πολλέ χρόνος. Α, είχαμε και τα πλαίσια αυτά του Brexit, οπότε η Ένωση ε, ε, έχει δεμένα τα χέρια, δεν μπορεί να σύναψε με κάποιους ε, εντάξει εταίρους με του οποίους συμμερίζονται κάποιες αξίες ε, όπως ο Καναδάς, πόσο πιο κοντά να είναι κάποιος. Όμως συνέχεια θα, θα, θα πρέπει να ταλαιπωρούμε και είπαμε τι γίνεται και με τα μεταλλαγμένα, στους δεν αρέσουν τα μεταλλαγμένα, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι από τον σχετικό κανονισμό κινδυνεύει καθόλου η Ευρώπη. και πάρα πολλοί συνάδελφοι όμως προσπαθούν με ιστερικό τρόπο να ασκήσουν αντιπολίτευση σε αυτήν την συμφωνία. Και αν κανείς ε, παρακολουθήσει την επιχειρηματολογία του εισηγητή, ε, τότε θα πρέπει ποτέ να μην συνάψουμε καμιά εμπορική συμφωνία. Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε 100% στεγανές εγγύσεις ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Ε, δεν είναι δυνατόν έτσι να συμφωνήσω μαζί του και εγώ και η πολιτική μου ομάδα. Δεν ξέρω τι θα πούμε ως ομάδα, αλλά δεν βλέπω να τον υποστηρίζουμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κατενμάκη, για την άλλη. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε και θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα διεθνούς εμπορίου και θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή πώς στην πράξη αυτή η συμφωνία, η οποία όντως μπορεί να χαρακτηριστεί σαν η καλύτερη που έχει ποτέ συναυθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός τρίτου κράτους. Στην πράξη αυτή η, η συμφωνία πώς θα είναι υποφιλής για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, πώς θα προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους αλλά και τις ε, δραστηριότητες. Δεν θέλω κενές ε, φράσεις και λόγια που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, πώς θα βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος μέσω αυτής της ε, συμφωνίας. Και μία επιπλέον ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε, έτσι κατάλαβα, ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει τους πιο, ε, τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες ε, γεωργικών προϊόντων. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά και πώς γίνεται. Και η τελευταία ερώτησή μου αφορά την προστασία των επενδύσεων. Καταλαβαίνω ότι αυτή η συμφωνία διασφαλίζει και προστατεύει τις επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως διασφαλίζονται και προστατεύονται και οι εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και το περιβάλλον και η ασφάλεια των τροφίμων και η δημόσια υγεία. Νομίζω ότι αυτές οι πτυχές είναι εξαιρετικά σημαντικές για μας. Μιλήσατε για αυτό το νέο σύστημα επίλυσης των διαφορών και προστασίας των επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι που υιοθετήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Καναδά, είτε ήταν πρωτοβουλία δική μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα επίλυσης των διαφορών και προστασίας των επενδύσεων. Από ό,τι είχα καταλάβει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα κράτος δικαίου, ένα συγκεκριμένο νομοθετικό σύστημα. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στον Καναδά, το γνωρίζω. Γιατί λοιπόν ε, απαιτείται ένα τέτοιο σύστημα το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε, δεν αρκούν τα δικαιοδοτικά όργανα στην κυριαρχία των ε, ευρωπαϊκών κρατών. Από τη στιγμή που μία ευρωπαϊκή επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, τηρεί πρότυπα ασφάλειας, δημόσιας υγείας, συνθήκων εργασίας για τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα βαίνουν καλά. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν παραβιάσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, δεν μπορεί να προσφύγει η επιχείρηση ή ο εργαζόμενος στα δικαστήρια είτε τη χώρα είτε στα διεθνή δικαστήρια. Θα ήθελα, αν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, να μου στείλετε μια γραπτή απάντηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ήμουνα στην Ίντα, που ήμουν ε, η συγγήτρια για την έκθεση αυτή. Και εκεί συζητήσαμε για το ΣΕΤΑ, αλλά αναβλήθηκε ε, τελικά η συνέχεια, γιατί παραμένουν ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με την συμφωνία αυτή. Σίγουρα είναι περίπλοκο το ζήτημα. Το ξέρουμε. Λοιπόν, χαίρομαι που η Ένβη θέλει να το συζητήσει και που θα μπορέσει να το συζητήσει για να αποφανθεί, όπως επίσης και η Επιτροπή Απασχόλησης και ίντα και οι μεταφορές. Σήμερα Πολλές ε, οργανώσεις έχουν ε, ζητήσει να εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Έχουμε όμως την αίσθηση, και ο κόσμος έχει την αίσθηση, ότι είναι μια συμφωνία η οποία συμφωνείται χωρίς αυτόν. Γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε η συζήτηση να γίνει για όλα τα πολύπλοκα ζητήματα αυτής της έκθεσης και για την κυρία Γκέρλινγκ. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί λέει κύριε Γκέλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά τη. Ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την εξουσία να ελέγχει. Πώ θα το κάνει αυτό, αν δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει αυτή τη τόσο μεγάλη συμφωνία με τόσο τεράστιε επιπτώσει. Ο συνάδελφο Στά έκανε έκκληση για το τι θα γίνει με την Joint αυτή Committee, με τη μεικτή αυτή επιτροπή που θα μπορεί να αλλάζει πράγματα και να έχει το πάνω χέρι, πάνω και από την νομοθεσία, την εθνική. Εμείς πρέπει να πείσουμε, να πείσουμε και να πιέσουμε για δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό το σύστημα του επενδυτικού δικαστηρίου δεν ε, λειτουργεί. Δεν ε, βοηθάει και πολύ, δεν είναι και πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε πριν εδώ είδαμε παραδείγματα. Γιατί να μην μπορούμε με το ήδη υπάρχον δικαστικό σύστημα στην Ευρώπη να διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Υπόθηκαν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων, οι ορμόνες ανάπτυξης, θυροειδής, ένα σωρό προβλήματα και υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για το τι τελικά θα προσφέρει η ΣΕΤΑ. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ερώτημα. Εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Στη ΣΕΤΑ ε, μιλάμε επίσης για υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για φυσιοθεραπεία, παραϊατρικές υπηρεσίες. Πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για όλους. Λοιπόν, όλα αυτά να τα κοιτάξουμε καλά και να τα ερευνήσουμε καλά. Αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το να έχουμε μία εμπορική συμφωνία είναι φυσικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αν ασχολείται μόνο με το εμπόριο. Ναι, αλλά πώς με το εμπόριο και πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν θα είναι καλό για το περιβάλλον ή όχι. Και να έχουμε και ισότιμες συνθήκες για όλα. Ενώ τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι μειώνονται οι προδιαγραφές για τον ε, παραγωγό κάνει το ίδιο, γιατί αν οι προδιαγραφές είναι υψηλές παντού, τότε είναι τάξη και για αυτόν. Το πρόβλημα του είναι όταν δεν είναι ισότιμες οι προδιαγραφές και είναι αλλού υψηλές και αλλού χαμηλές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Κοντά, εκ μέρου του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή για τη ΣΕΤΑ είναι μια εξαίρετη ευκαιρία να δείξουμε τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μάλλον το πόσο άχρηστο είναι. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριο Στάς μας παρουσίασε διάφορες ε, συνθέσεις που είναι σαφέστατες. Η μεικτή Επιτροπή μα το είπε, μπορεί να τροποποιήσει τα νομοθετικά κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί να μπορούν οι ευρωβουλευτέ να πούνε τίποτα. Μα τα παραρτήματα που μπορεί να τροποποιήσει η Μικτή αυτή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά, γιατί αναφέρει ποια είναι τα παρασυντοκτόνα που επιτρέπονται, κάποιε ουσίες στα τρόφιμα ή με ποιο τρόπο βάζουμε ετικέτε, τι λένε ετικέτε στα τρόφιμα. Συνεπώ, η συμφωνία αυτή καταδεικνύει πόσο περιφρονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τους εκλεγμένους της και λειτουργεί αλλά καρτ. Γίνονται διαπραγματεύσει σε μικρέ επιτροπέ, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει έλεγχο και δεν υπάρχει και αντιπαράθεση. Θα έπρεπε η συμφωνία αυτή, αν μη τι άλλο, να προβλέπει προσφυγή σε περίπτωση κατεξοδότηση πράξεων, όπου να έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ούτε καν αυτό προσπαθεί. Και μάλιστα εμείς που είμαστε μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε δικαίωμα να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που φαντάζομαι ότι δεν θα μας λάβει υπόψη όπως έγινε και με την γνωμοδότησή μας για το TTIP. Τα φυτογενομικά μέτρα όμως είναι ζωτική σημασία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε λοιπόν, και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι η ΣΕΤΑ είναι ό,τι καλύτερο ω εμπορική συμφωνία, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η καλύτερη συμφωνία είναι μια συμφωνία όπου δεν έχουν δικαίωμα λόγου οι ευρωβουλευτέ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ο κύριο Λίζε τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, να σας πω κάτι διαδικαστικό. Εάν υπάρχει πίεση χρόνου, σε σχέση με το πότε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτήν την έκθεση, ε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Από πλευρά δική μα, γιατί οι άλλε επιτροπέ νομίζω ότι προχωρούν όσο ταχεία πρέπει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ρίχνουμε το φταίξιμο σε άλλου. Πάντω, γενικώ η εντύπωση μου είναι από τις επαφές που είχα στην εκλογική μου περιφέρεια ότι η κοινή γνώμη θεωρεί ότι σε επόμενες έξι εβδομάδες κάτι θα πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων ε, υπάρχει γενική συνένεση υπέρ και ε, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί κάποιοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α, ας πούμε, το Κοινοβούλιο της Βαλανίας θέλουν να δυναμητήσουν αυτή την πορεία, αυτή τη συμφωνία. Ε, γι' αυτό και κόλλησε η πρόοδος των πραγμάτων. Νομίζω ότι τα θέματα έχουν ξεκαθαριστεί και για το κρέας ο Καναδάς συνεφώνησε, φώνησε δέχτηκε αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξαγωγές Μα αν κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν έχουν όλα ρυθμιστεί στο 100% μα για καθίστε, για σκεφτείτε. Αν δεν υπήρχε η ΣΥΤΑ θα ήταν πράγματα πολύ χειρότερα. Δεν θα είχε τίποτα λυθεί. Μα είναι δυνατόν εμείς να έχουμε πάντοτε το πάνω χέρι. Έτσι κι αλλιώς οι επαφές και τα προβλήματα αυτά συνεχίσουν από διάφορους φορείς να συζητώνται. Οι δε σοσιαλδημοκράτες στην ε, Γερμανία με τον κύριο Γκάμπριλ των εξωτερικών και ίσως ε, τον κύριο Στάνιμαγερ τον αυριανό ενδεχομένως ε, πρόεδρο. Είπε ότι πρόκειται για ε, ότι, ότι η είναι καλή συμφωνία και τι κακή. Τι δεν καταλαβαίνω για τα λένε όλα αυτά. Έχει παγώσει το TTIP. Όμως το γεγονός ότι λέμε ότι η ΣΕΤΑ είναι μια καλή συμφωνία. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο παραπάνω με τους Καναδούς ομολογούς μας. Εγώ μίλησα με τον ε, Καναδό πρέσβη και πολλά πράγματα από αυτά που δεν δέχονται οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Καναδάς τα δέχτηκε στη συμφωνία μαζί μας. Καταρχήν ο Καναδάς δεν θέλει να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θέλει λοιπόν να έχει πιο ισορροπημένες εμπορικές τέχεις. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρόλος εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι καθοριστικός. Το ερώτημα είναι με ποιον άλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία. Ξέρουμε ότι η χώρα αυτή, ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία κυβερνάται από μια φιλελεύθερη κεντροαριστερή κυβέρνηση και με ποιον άλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρόμοια, να συνάψουμε μια παρόμοια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τέτοιες ευκαιρίες. Η Ευρώπη χρειάζεται ε, αυτές τις δυνατότητες, χρειάζεται την προστασία των προτύπων για τους καταναλωτές μας και για τους ε, εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ακούω τους πράσινους έχω την εντύπωση, και εδώ αναφέρομαι και στον κύριο Στάς, και σε όλο το φάσμα των κριτικών που ακούγονται από την άκρα αριστερά ως την άκρα δεξιά. Ελπίζω ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα τεθούν υπέρ αυτής της πολύ προοδευτικής συμφωνίας, η οποία πραγματικά προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Πόρετ. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Φορίντσα. Ευχαριστούμε και για την ε, έκθεση. Θα μπορούσα να πω ότι την συμφωνία ΣΕΤΑ την χαρακτηρίζει ως την καλύτερη δυνατή από πλευρά μας ε, συμφωνία. Από την άλλη μεριά όμως δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό. Πάντως θα πρέπει να γίνει αυτή η ζήτηση πλευρά μας, γιατί αυτό το οποίο θέλαμε είναι να συνδεθεί αυτή η συμφωνία και να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε, διότι Υπάρχουν τα θέματα για το περιβάλλον, για την ενέργεια, για την ε, δημόσια υγεία που είναι δικές μας αρμοδιότητες. Και ρυθμίσεις ε, ε, αυτές δεν είναι καθόλου ευχάριστες, αλλά θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συζητήσει τη Συμφωνία ΣΕΤΑ και αυτό να γίνει επιγόντως. νομίζω ότι δεν έχουν ζητηθεί. Δεν συζητούνται αρκετά οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται. Ακριβώς αυτό σα τονίζω ότι αναδύεται από αυτό το, το, το, σχέδιο του κειμένου ε, και από τα όσα έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντως όσον αφορά την ουσία της συμφωνίας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που η ουσία της συμφωνίας, όπως όλες οι συμφωνίες οι εμπορικές μιας γενιάς, δεν καλύπτει τα θέματα των δασμών, αλλά καλύπτει τα θέματα των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Οπότε έχουμε τώρα αυτά τα ε, πρότυπα για ευαίσθητα εμπόρια και, εμπόρια και για εμπορεύματα μάλλον και για θέματα επίσης ευαίσθητα όπως το περιβάλλον και δημόσια υγεία. Εγώ να σα ρωτήσω τα εξή. Αφού κατηγορώντα κάτι θα πρέπει να γίνει για το κλίμα, θα πρέπει πολιτικά να δω κάποιε λύσει και αφού η ΣΕΤΑ δεν καλύπτει αυτές τι ε, ανησυχίε. και στο προήμιο της συνθήκη δεν γίνεται παραπομπή στη Συμφωνία των Παρισίων, ούτε στην μείωση των βλαπτικών αερίων για το θερμοθερμοκηπίο. Στο τέταρτο κεφάλαιο εκεί. Ε, επίσης δεν αναφέρεται ε, τίποτα στο, στο βασικό ε, σημείο του κειμένου για το περιβάλλον. Επίσης, κεφάλαιο 22 και 24. Ούτε εκεί οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον είναι νομικά δεσμευτικές. Άρα λέμε για το τι γίνεται με το εμπόριο και τι γίνεται με τις επενδύσεις, αλλά δεν προβλέπεται ε, σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες κανός είδους κύρωση αν γίνει παραβίαση των περιβαλλοντικών διατάξεων. Άρα θα έπρεπε νομίζω η πολιτική μας να διέπεται από περισσότερη μέρη για το περιβάλλον και για την ενέργεια επίσης. Για πέστε μου, καλύπτει η τσέτα το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο. Καλύπτονται αυτά ως εμπορεύματα. Αυτά προβλέπεται να εισάγονται χωρίς δασμούς επίσης. Κάτι άλλο. Όσον αφορά την ε, εναρμόνιση, γίνει η εναρμόνιση προς τα κάτω. Τα είπαμε αυτό από το Σεπτέμβριο του 2014. Και είπαμε ότι θα πρέπει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων να είχαν πει να εξαιρεθεί το ε, πετρέλαιο, αλλά επίσης και τα ορυκτά καύσιμα. Όμως πρέπει να πάμε σε βιώσιμες, σε ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και έτσι να μην έχουμε εκπομπές διευθύντου του άνθρακος. Τώρα ποια είναι η σχέση του Τσέτα και των μεταλλαγμένων ιδίως όσον την ειδικετοθεσία. Θα πρέπει να, δούμε τι γίνεται για, όσον αφορά την προέλευση των ε, τροφίμων στην Ευρώπη υπάρχουν απαγορεύσει σε σχέση με τα μεταλλαγμένα. Γι' αυτό και το 2003 έγινε η σχετική ρύθμιση όσον αφορά τα δικά μας μεταλλαγμένα. Όμως, με τώρα με την ΣΕΝΤΑ, όσον αφορά τα μεταλλαγμένα, ασκείται πίεση στην Ευρώπη. Και τώρα δεν υπάρχει μία επιστημονική προσέλευση προ, είναι προσέγγιση τέτοια. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να προστατευτεί η υγεία ανθρώπων και ζώων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικά. Και ε, ευτυχώς ε, μετακινήθηκε στην Ίντα η ημέρα της ε, ψηφοφορίας και έτσι ελπίζω να μπορέσουμε εμείς να γνωμοδοτήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Κυρία Γκροστέτ, έχετε το λόγο. Προσπαθήσω να είμαι γρήγορη και σύντομη, Πρόεδρε. Διαβάζοντας αυτή τη συμφωνία διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι τόσο τρομερό όπως το περιγράφουν το κείμενο αυτό κάποιοι. Ας κοιτάξουμε αυτή τη συμφωνία με ρεαλισμό και Καταρχήν χαίρομαι για το άρθρο 8.9, το τμήμα Δέλτα αναφέρεται στην ε, δυνατότητα που έχουν τα διάφορα μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη, να υλοποιήσουν για θέματα ασφάλειας, προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώματα, τα οποία παραμένουν κυρίαρχα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κάποιες άλλες διαφορές σε θέματα επενδύσεων είτε κερδών για τους επενδυτές. Με μεγάλη επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον είδα και τα θέματα των δικαιωμάτων όσον αφορά την αξιολόγηση των προϊόντων που αφορούν την υγεία καθώς και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας. Όσον αφορά την έρευνα και θέματα συνεργασίας σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή πώς αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να πλήξει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και της αντίστοιχης υπηρεσίας ε, του Καναδά. Για το θέμα των φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει προβλέψει όσον αφορά τις διατάξεις για τα άρθρα 2027 και 2028. 28. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις για την τιμή αυτών των φαρμάκων. Τι θεωρεί η Επιτροπή ότι θα είναι η συνέπεια επί των τιμών σημαντική ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάτσο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να αντιδράσω σε κάτι που άκουσα νωρίτερα. Εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε οι επαγγελματικές ιδεολογικές συζητήσεις. Ο κύριος Λίζη για πρώτη φορά έθεσε πολιτικά το ζήτημα όταν επιτέθηκε στους πράσινους και τους ε, κατηγόρησε για τη συνεργασία τους με κάποιους ευρωβουλευτές. Θα μπορούσα να κάνω και εγώ αντίστοιχες παρατηρήσεις για τους χριστιανοδημοκράτες, για το ΕΛΚ, αλλά δεν θα το κάνω. Έχω μια ερώτηση. Το TTIP έχει παγώσει προς το παρόν. Τι θα γίνει αν το TTIP δεν γίνει ποτέ πραγματικότητα. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιήσουν τη συμφωνία ΣΕΤΑ θηγατρικές αμερικανικές δηλαδή μεσολαβήσουν ώστε να πετύχει η Αμερική αυτά που ήθελε να πετύχει με το TTIP. Οι εμπορικές μας σχέσεις με τον Καναδά είναι περιορισμένες. Τώρα, συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι πρέπει να αναλύσουμε καλά αυτή τη συμφωνία και πρέπει να έχουμε μια θετική στάση, είπαν κάποιοι. Εγώ συμφωνώ για το ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και η προσέγγιση μου είναι θετική να διατηρήσουμε τις δικές μας προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και έχω και θετική προσέγγιση και όσον αφορά την εθνική μας κυριαρχία. Δηλαδή με άλλα λόγια, αν μια εκλεγμένη κυβέρνηση εκπονήσει έναν κανονισμό, μια νομοθεσία, δεν είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να προσφύγει σε βάρος της, σε βάρος της ε, χώρας αυτής της κυρίαρχης και αυτό κάνει το σύστημα διατησίας που προβλέπεται στη ΣΕΤΑ. Θα θυμόσαστε ότι και στον ΟΣΑ έχει υπάρξει συμφωνία για έναν μηχανισμό πολυμερή προστασία των ε, επενδυτών. Δεν έγινε πολυμερός αυτό και τώρα η προσπάθεια είναι να γίνει διμερός. Ελπίζω να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Κονέτσκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ προηγούμενοι ομιλητές ε, ανέφεραν τα περισσότερα από αυτά που θα ήθελα να πω, το θέμα της ασάφειας που υπάρχει για το περιβάλλον, παραδείγματο χάρη, το θέμα της διατησίας, η ρύθμιση, παραδείγματο χάρη κάποιων κρατικών προμηθειών, οι κανόνες, η δυνατότητα των κυβερνήσεων να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, Πρέπει να θέσουμε πολύ φιλόδοξους περιβαλλοντολογικούς στόχους στην πολιτική μας. Και η συμφωνία αυτή, όπως την διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι λίγο αντίθετη με αυτό που προσπαθούμε εμείς εδώ τόσα χρόνια να πετύχουμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να ρυθμίσουν από μόνες τους αυτά που επιθυμούν όταν πρόκειται για πολύ αυστηρούς κανόνες που αφορούν το περιβάλλον. Δεν μπορεί να τα καταστρέψουμε αυτά και να τα εξαλείψουμε. Εδώ κινδυνεύει αυτή η πολιτική. Υπάρχει ένα κεφάλαιο, παραδείγματο χάρη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για κενά λόγια. Δεν πρόκειται για δεσμευτικές προτάσεις. Και αυτό που με ξαφνιάζει ιδιαίτερα είναι ότι η Συμφωνία ΣΕΤΑ αφορά και το νερό σαν να επρόκειτο για ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν συναλλαγών. Το νερό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα. Δηλαδή η πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι καθοριστικό για τους πολίτες μας και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το νερό θα γίνει προϊόν εμπορίας. Οι οικονομικές σας αναλύσεις μας δείχνουν ότι μόνο 1% αυτών των διευθετήσεων αφορούν την εμπορική αξία και το κέρδος. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ούτε το περιβάλλον, ούτε την προστασία της υγείας και όλα αυτά φαίνεται δεν σας αφορούν. Αυτό που διαπραγματευτήκατε και το αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής είναι για μας απαράδεκτο. Και ε, κύριε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε δεν προχωρήσουμε τη συμφωνία με τον Καναδά, τότε τι. Αλλά το είπε και η κυρία Κροστέτ για τα άρθρα 8, 9, 10. Όμως έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Επιτροπή. Η Ολλανδία λέει ότι κοιτάμε περισσότερο τους δασμούς και λιγότερο τα εμπορικά μέτρα. Η μελλοντική συμφωνία έχει συμφωνηθεί για να αναγνωριστούν αμοιβαία οι προδιαγραφές και τα προϊόντα της άλλης χώρας που είναι χαμηλότερων προδιαγραφών να μπορούν να μπουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέγονται στην Ολλανδία. Και είμαι και εγώ επικριτική. Έχω πει ότι πρέπει να κοιτάξουμε, είμαι υπέρ της συμφωνίας, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μήπως υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι θα πληγούν αλλά με το 8, 9 και 19 τα άρθρα αυτά νομίζω είμαστε σε ισότιμους όρους. Είναι έτσι ή όχι. Είναι ερώτηση αυτή που κάνα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να απαντήσουμε στις επικριτικές. Ακούω και τους αγρότες στη χώρα μου που λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες από την Ευρώπη και θα υπάρξουν και άλλες διεθνείς συμφωνίες που να μην έχουν καν ε, ψηφιστεί από τους Ευρωπαίους. Είναι και αυτό ένα επιχείρημα που λένε οι αγρότες στη χώρα μου και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρόεδρος, καλώς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στην πληθώρα των ερωτήσεων. Έχουμε διερμηνία για λιγότερο από 10 λεπτά. Μετά θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλέ ήταν οι ερωτήσει να τις ομαδοποιήσουμε και να τις απαντήσουμε. Πολλές ερωτήσεις είχαμε όσον αφορά τις αρμοδιότητες της κοινή επιτροπής. Ποιες είναι και ποιες δεν είναι. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είναι μια εξωτερική ανεξάρτητη επιτροπή. Συναποτελείται από Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά τους, συμβαλωμένους. Και για να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Επιτροπής είναι δυνατόν μόνο εάν συμφωνήσει το Συμβούλιο σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχυρή διαδικασία. Δεν μπορεί να τροποποιήσει αυτή την επιτροπή το ε, κείμενο της συμφωνίας. Μόνο κάποια παραρτήματα, όπως αναφέρατε κάποιοι από εσάς και οποιαδήποτε αλλαγή της συνθήκη θα πρέπει να ακολουθήσει την πλήρη διαδικασία με συμμετοχή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Μπορεί μόνο να τροποποιήσει αυτή η επιτροπή για το SPS κάποια παραρτήματα. Και αυτή η απόφαση για τα φυτοϊγειονομικά θα πρέπει να ακολουθήσει τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι παρεκκλήσεις δεν προβλέπονται. Επίσης θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της πρόληψης και αυτά τα οποία ανέφεραν πολλοί ε, συμβουλέ, για διάφορε βουλευτές για τα MRL. Δεν μπορούν να γίνουν επομένω άλλε αλλαγέ από τα μέλη τη ε, Γενικής επιτροπή, όσον αφορά τα ε, ντομοκτώνα, ε, τα παρασυτοκτώνα και τις συναφεί ουσίε. Σημαντικό αυτό να αναφερθεί. Επίσης οποιαδήποτε απόφαση για ισοδυναμία Μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν ενδελεγού αναλύσεω. Δηλαδή να έχουμε κάποια τέτοια μέτρα για τα φυτογειονομικά, αυτά ε, ε, διέπονται από αμοιβιότητα, από αντιστοιχεία ή κάποια, κάποια άλλα μέτρα τα οποία ε, έχουν προταθεί. Οπότε ό,τι και να αποφασιστεί συνάδει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Επιτροπή. Είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την ε, μελετά η αρμόδια επιτροπή και κατόπιν ε, αποφασίζει η κοινή επιτροπή. Αυτά είναι δικές μας ε, διαδικασίες, αλλά και ο Καναδάς έχει αντίστοιχες. Τίποτα στην συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει τα πρότυπα για τα είδη διατροφής ούτε για τα μεταλλαγμένα, ούτε για τις ορμόνες. Οπότε, ό,τι εισάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από αυτούς τους κανόνες. Κάποιο κατάρριξη δασμών ή ποσοστώσεων που προβλέπονται υπέρ του Καναδά στη ΣΥΤΑ και οποιαδήποτε ε, προϊόντα καναδικά που διέπονται από αυτές τις ποσοστώσεις θα πρέπει να συνάδουν προς την νομοθεσία μας για τα ίδια διατροφής. Δεν παρακάπτεται η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό το ορίζει η συμφωνία, αλλά όχι μόνο. Και στο κοινό έγγραφο ερμηνεία της συνθήκης που έχει δυσμευτική ισχύ σύμφωνα και με το άρθρο 31 Συνδίκη της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνδικών. Οπότε και σε αυτό το κείμενο τονίζεται σαφώς το ζήτημα και γίνονται και παραπομπές στο κείμενο, στο σώμα της συνθήκης. Για όλα αυτά που είπαμε και για τα πρότυπα που αφορούν τα τρόφιμα. Τώρα αυτή η αρχή της σοφροσύνης, της πρόληψης που προβλέπεται από τη Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά και δεν μπορεί να αλλοιωθεί από την ΣΥΤΑ. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ζωητή παραπομπή σε αυτή την αρχή από τη ΣΥΤΑ, τότε κατησχεί το κοινωτικό δίκαιο και για τα μεταλλαγμένα πρόσωπα το περιβάλλον. Τι δεσμεύσει έχουν αλληλευθεί. Εκεί που υπάρχουν θέματα απασχόλησης και εμπορίου στα σχετικά κεφάλαια η Επιτροπή θεώρησε ότι ό,τι δεσμεύσει προβλέπονται εκεί έχουν δεσμευτική ισχύ. Οπότε τα κρατημέλη θα πρέπει να λογοδοτήσουν έναντι των υποσχεσιών του. Και για την απασχόληση, για πρώτη φορά ο Καναδάς σε μια εμπορική συμφωνία έχει δεσμευτεί σε αυτά, για αυτά τα σημεία σε σχέση με τις συμφωνίες με το Εθνές Γραφείο Εργασίας γιατί δεν έχει γίνει η κύρωση τεσσάρων από τις οκτώ συμβάσεις του ILO, του Ιθνούς Γραφείου Εργασίας. Αλλά τρεις της εκκύρωσης από το πρόσθεσμα διαπραγματεύσεις. Ακόμα εκκρεμία η μία για τις συλλογικές συμβάσεις και η κυβέρνηση Τριντό άρχισε αυτή τη ε, διαδικασία κύρωσης, οπότε γίνονται διαπραγματεύσεις και αυτές μπορούν να έχουν ε, θετικές επιπτώσεις, τόσο ώστε να γίνει κύρωση των ε, όσων προβλέπει ο ILO. Και έτσι για το περιβάλλον έχουμε διάφορες πολυμερείς συμφωνίες, αλλά και τη συμφωνία των Παρισίων που πάει προς κύρωση. Όντως δεν αναφέρεται ρητός στο κείμενο της ε, ΣΥΤΑ. Αλλά διαπραγματεύσει για το κείμενο της ΣΥΤΑ ολοκληρώθηκαν πριν ε, ολοκληρωθεί η σύνοδος των ε, και υπογραφή σχετική συνθήκη. Όμως είναι σαφής η πρόθεση των ε, συμβαλωμένων. Αυτό το αναφέρει και αυτό το ερμηνευτικό κείμενο. Ότι θα ληφθεί υπόψη η Συμφωνία των Παρισίων. Πολύ σημαντικό αυτό. Πέραν του του πάντως έχουμε κάποιες ε, διατάξεις που αναφέρονται στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, στην κοινωνική ευθύνη Και τελευταίο και σημαντικό, τα σχετικά κεφάλαια προβλέπουν για κάποιους μηχανισμούς μηχανισμούς κάποια κρατημέλη. Ε, φρόντισαν τους ώστε να υπάρχουν και αυτοί οι μηχανισμοί εφαρμογής και όχι μόνο οι, α, οι δεσμεύσεις. Πέραν λοιπόν των α, ε, κεφαλαίων αυτών Γενικότερα, η ΣΥΤΑ έχει την ίδια προσέγγιση όπως όλες οι εμπορικές συμφωνίες. Πρώτα πρώτα υπάρχει μια διαβούλευση, δεν υπάρχει κάποιο θέμα ε, και ο ένας συμβαλόμενος το λέει στον αντισυμβαλόμενο και ξεκινάει η διαβούλευση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αν ε, αυτή η πρώτη κίνηση δεν λύσει το πρόβλημα, τότε πάει στο πάνελ των ανεξαρτήτων εμπειρογνωμών και επίσης υπάρχει και η Επιτροπή του Εμπορίου και της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπου και το θέμα συζητείται και αυτό το πάνελ θα πρέπει να δημοσιοποιήσει μια έκθεση πάνω στο πρόβλημα και αν δεν βρεθεί κάποια λύση τότε προβλέπονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί στα σχετικά κεφάλαια ούτως ώστε να γίνει επίλυση των διαφορών. Ναι, οπότε αυτές οι δεσμεύσεις είναι δεσμευτικές. Τώρα όσον αφορά την νομοθετική συνεργασία, σα τονίζω ότι αυτή η συνεργασία προβλέπεται ρητό στο 21 παράγραφο 2. Είναι εκουσία, ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών. Αυτό αφορά δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι η ρύθμιση. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσει η διερμηνία, όπως προβλέπετε. Ευχαριστώ. Of agricultural products, um, I mean, yes, the EU opens its market on, for certain um, certain areas, uh, certain products where this is of the interest of Canada, but at the same time, the EU has